Λοιπόν, ε, σήμερα είναι η 37η ημέρα των κινητοποίησεών μα, ένδειξη διαμαρτυρία για τη μονομερή επιβολή άδικης, αδικών, άδικων συνθήκων εργασία για του διερμηνεί από πλευρά τη Δίκη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και γι' αυτό με τα λύπη μα σα ενημερώνουμε ότι η διερμηνία θα σταματήσει ακριβώ την προβλεπόμενη ώρα. Ευχαριστούμε. Ε, λοιπόν, ο χρόνος μας είναι περιορισμένος και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Μπετίνα Γιάκοψον. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω την έκθεσή μου για την ενίσχυση της ικανότητας των διεθνών δυνάμων ασφαλείας στην Ιγυρία και στο Μάλι. Είναι δύο χώρες ε, στην Αφρική, νεαρές δημοκρατίες με αδύναμα διοικητικά συστήματα. Το 2007 η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, εκπώνησε ένα πρόγραμμα στην προϋπόθεση ότι η ανάπτυξη και η ασφάλεια αλληλοσυμπληρώνονται και τα προβλήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε περιφερειακό επίπεδο. Ε, υπάρχουν πολλές αποστολές καθώς και στρατιωτικές επιχειρήσεις αποστολές πολιτικής φύσης και στρατιωτικές επιχειρήσεως στο πλαίσιο της ατυχής της Ευρωπαϊκής ε, ε, Ένωσης προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απειλές και να εξασφαλίσουν την, τις συνθήκες ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ενισχύσει την ικανότητα των διεθνών δυνάμεων που είναι υπεύθυνε για την ασφάλεια παράγοντας ε, κατάλληλη κατάρτιση και εξοπλισμό. Το Συμβούλιο ε, δηλώσε ότι θα ενισχύσει τις προσπάθειες αυτές ε, πάταξης του οργανωμένου εγκλήματος. Και υπήρξε μια διεύρυνση της ε, εντολής Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, όσον αφορά την καταπολέμηση αυτή του οργανωμένου εγκλήματος και τις πληροφορίες για την παράνομη μετανάστευση. Ε, επίσης υπάρχει προσπάθεια να στηριχθούν οι τοπικές αρχές όσον αφορά τη διατήρηση της δημοκρατικής τάξης και τις ε, δημιουργίες ε, μόνιμων συνθήκων ειρήνευσης στο Μαλί και ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας μέσω μιας προσπάθειας ενίσχυσης της διακυβέρνησης της χώρας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο <clears throat> έθεσε ε, στην διάθεση αυτών των επιχειρησιακών μονάδων ε, σημαντικά οικονομικά κονδύλια. Ο στόχος μας ήταν να εξετάσουμε πώς η UCAP αποστολή λειτουργήσε στις χώρες αυτές και πώς πέτυχε να ενισχύσει τις ικανότητες των δυνάμεων που είναι υπεύθυνε για την εσωτερική ασφάλεια των δύο χωρών. Εμείς ε, ε, για να το αξιολογήσουμε ε, θέσαμε δύο ερωτήματα κατά πόσο ήταν σωστή η εφαρμογή των GU CAPS και δεύτερον ενίσχυσαν οι αποστολές αυτές τη δυνατότητα, την ικανότητα των δυνάμεων ασφαλείας στην Ιγυρία και στο Μαλί. Αυτό το οποίο βρήκαμε ήταν το εξής. Καταλήξαμε συνολικά στο συμπέρασμα ότι οι αποστολές συνέβαλαν στην ενίσχυση της ικανότητας των δυνάμεων που είναι υπεύθυνε για την εσωτερική ασφάλεια, αλλά η διαδικασία επιβραδύνθηκε από τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν και από ε, ε, επιχειρησιακά προβλήματα. Και επιτρέψατε μου να αναφέρω ορισμένα από τα βασικά ευρήματα και συμπεράσματα στον έλεγχό μα. Η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα επηρεάστηκε αρνητικά από ένα συνδυασμό ε, θετίας δύο ετών, προβλημάτων προϋπολογισμού κλπ. Ε, η στελέχωση του προσωπικού δεν ε, είχε επαρκή καθοδήγηση και στην Ιγυρία ε, δεν ήταν επαρκής η εκπαίδευση των στελεχών σε ορισμένες ε, περιπτώσεις εφαρμόστηκαν διαδικασίες που ήταν, ε, δεν ήταν ενδεδειγμένες για τις συνθήκες που ήσχαν στην ε, περιοχή αυτή. Και θα ήθελα να σας δώσω δύο παραδείγματα. Επειδή η αποστολή συστάθηκε ταχύτατα, οι λογιστικές διευθετήσεις δεν υπήρχαν ευθύ εξ αρχής και χρειάστηκαν 18 μήνες για την αποστολή προκειμένου να συγκροτηθεί η οντότητα. ρε επικεφαλής των αποστολών έπρεπε να υπογράψουν όλα τα έγγραφα με το δικό τους όνομα ε, και γι' αυτό έφεραν αυτή την ε, νομική και οικονομική ευθύνη. Επιπρόσθετα η αποστολή δεν είχε δικό της προπολογισμό για την φάση εκκίνησης, άρα είχε μια βραδία εκκίνηση ως φορά την διεξαγωγή δραστηριοτήτων, γιατί είχαν πενιχρή ε, διοικητική και λογιστική υποστήριξη από τις Βρυξέλλες. Στην Ιγυρία αυτό δεν περιορίστηκε μόνο στην αρχική φάση, αλλά συνέχισε και τα επόμενα χρόνια διεξαγωγή των επιχειρήσεων. Ε, στο, στα προγράμματα τα οποία ελέγξαμε υπήρξαν καθυστερήσεις ε, στα ε, προγράμματα κατάρτισης. Σε πέντε περιπτώσεις το στέλεχος είχε υποβάλει κάποιες εκτίσεις για τον εξοπλισμό, αλλά τελικά είχαν εγκαταλείψει τη θέση εργασία τους πριν φτάσει ο εξοπλισμό αυτό. Επίση, η κατάρτιση ήταν ατελή, πράγμα που οδήγησε καθυστερήσεις <clears throat> στις ε, αποσταλές αυτές. Επίσης, ε, πολλά από τα στελέχη τα οποία ήταν υπεύθυνα για την προπαρασκευή των τεχνικών προδιαγραφών δεν είχαν ε, σαφή γνώση των διαδικασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κανόνων. Αυτό οδήγησε επίσης σε καθυστερήσει διαδικασίες προμήθειας και οδήγησε σε ακυρώσει των συμβάσεων. Ένα άλλο παράδειγμα αφορά την κατάρτιση που δόθηκε στι δυνάμει εσωτερική ασφαλεία. Λόγω ε, προβλημάτων στη διοίκηση, οι αποστολέ δεν ήταν σε θέση να παράσχουν πλήρη τεκμηρίωση για τα μισά προγράμματα κατάρτιση, όπως για παράδειγμα τι αξιολογήσει κλπ. εκ μέρου των συμμετεχόντων. Η αποστολή στο Μαλί είχε καλύτερα αποτελέσματα εδώ. Τώρα, όσον αφορά το τοπικό κέντρο στην Ιγυρία, παρόλο που η αποστολή είχε παράσχει τον εξοπλισμό στο κέντρο αυτό, δεν ήταν λειτουργικό γιατί δεν υπήρχαν καθίσματα, έλειπαν τα τρεπάζια, ε, τα τραπέζια, συγγνώμη, και ο κλιματισμός δεν λειτουργούσαν. Άρα οι αποδέκτες ε, δεν ε, μας έδειξαν τους υπολογιστές που είχαν λάβει, εκτυπωτές δεν λειτουργούσαν και ο εξοπλισμός για τις ραδιοπικοινωνίες δεν λειτουργούσε. Δύο οχήματα τα οποία θα έπρεπε να είναι στη διάθεση του κέντρου προκειμένου να ανταποκρίνεται ταχαίως έκτακτες ανάγκες ποτέ δεν είχαν χρησιμοποιηθεί. Ένα από αυτά είχε βλάβες που δεν μπορούσαν να επισκευαστούν ήδη από το 2014. Άρα λοιπόν βρήκαμε ότι οι αποστολές προσπαθούσαν να καθαστήσουν ε, βιώσιμες αποστολές χωρίς επιτυχία παρά τη θετική ε, άποψη των αποστολών οι κυβερνήσεις στις δύο χώρες δεν ήταν πάντοτε διατεθειμένες να εγκρίνουν την κατάλληλη νομοθεσία και να περάσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις ε, προκειμένου να είναι βιώσιμα τα αποτελέσματα της ανάπτυξης ικανοτήτων. Στο Μαλί η κατάσταση επιδεινώθηκε και από την έλλειψη πολιτικής σταθερότητας και από οργανωτικά ελλείμματα σε κυβερνητικό επίπεδο. Αυτό υπονόμησε τις προσπάθειες των αποστολών να καταστήσουν τα αποτελέσματα δραστηριοτήτων τους βιώσιμα. Ωστόσο, οι αποστολές ήταν επίσης υπεύθυνε για τις δικές τους αδυναμίες όσον αφορά την εξασφάλιση της βιωσιμότητας. Για παράδειγμα, η αποστολή της Νιγηρίας δεν μπόρεσε να ελέγξει πώς οι γνώσεις ε, που ε, κομίστηκαν στα, ε, που, που, στη, που, που, που αποκτήθηκαν συγγνώμη, στην κατάρτιση τελικά αξιοποιήθηκαν από τους συμμετέχοντες. Δεν υπήρχαν στοιχεία κατά πόσο τα μαθήματα αυτά είχαν ολοκληρωθεί και κατά πόσο οι συμμετέχοντες εκπαιδευόμενοι είχαν μπορέσει να εφαρμόσουν τις γνώσεις που απέκτησαν. Ε, τώρα, πιο θεραντικό είναι το εξή Όσον αφορά την, ε, τους εκπαιδευόμενους, στην, ε, για τον εξοπλισμό στην Ιγυρία και το Μαλί, η συνολική αξιολόγηση δραστηριοτήτων αποστολών ήταν θετική. Οι ενεχόμενοι εκτίμησαν θετικά τη δυνατότητα του προσωπικού των αποστολών να τους παράσχουν συμβουλές, πράγμα που δεν μπορούσε να γίνει στη βάση των εθνικών πηγών. Στην Ιγυρία οι δυνάμεις ασφαλείας και οι κυβερνήσεις επεσήμεναν την αξία της ε, μόνιμης παρουσίας των αποστολών σε σύγκριση με άλλους δωρητές. Και οι δύο αποστολές επίσης παρήχαν πληροφορίες και συμβουλές σε υποστήριξη των άλλων εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ε, ευρύτερων δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών μελών. Για παράδειγμα, οι αποστολές συνέβαλαν στο σχεδιασμό του, Ευρωπαϊκού, του κατασπιτεύματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αφρική σε σχέση με τις ε, μεταναστευτικές ροές και ε, χαρτογράφησαν κάποιες σε σχέση ε, με την μετανάστευση. Οι δωρητές επίσης ε, τόνισαν το σημαντικό ρόλο και των δύο αποστολών στο συντονισμό των δραστηριοτήτων στον τομέα ασφαλείας. Και δύο αποστολές σύστησαν σώματα προκειμένου να βελτιώσουν το συντονισμό με τις εθνικές αρχές ε, κάτι που στην αρχή δημιούργησε κάποια προβλήματα, αλλά τελικά απέβη, ετελεσφόρησε. Επίσης, ενέκριναν κάποιου μηχανισμούς για το συντονισμό και τη συνεργασία με άλλου ε, δωρητές. Στη βάση αυτού του ελέγχου, η οι που διατυπώνουμε είναι εξή. Το ελεγκτικό συνέδριο απευθύνει τη σύσταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα προκειμένου να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των αποστολών ε, την κάλυψη και τη στελέχωση του προσωπικού, ε, την ε, αποδέσμευση κονδυλίων και επίσης τη δημιουργία μιας στρατηγικής εξόδου από τα προγράμματα, να αυξήσει την βιωσιμότητα και να βελτιώσει δείκτες όσον αφορά την παρακολούθηση και την αξιολόγηση. Η Επιτροπή και η ΕΕΣ αποδέχτηκαν όλες τις στάσεις μας στις εκθέσεις ελέγχου και αναμένω την εφαρμογή αυτών των συστάσεων εις όφελος της ε, κατάστασης εσωτερικής ασφάλειας στην περιοχή καθώς και στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι ευτυχής να απαντήσω τα ερωτήματά σας. Ευχαριστώ. Okay. Uh, thank you. Σας ευχαριστώ κυρία Γιάκοψεν. Okay. Και τώρα θα περάσουμε στην, στο κομμάτι με τις ερωτήσεις και απαντήσεις. Ο κύριος Γκάλερτ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση και πιστεύω ότι εδώ υπάρχουν δύο σφαίρες ε, που θα πρέπει να διατυπωθούν ε, τα ερωτήματα και να δοθούν οι απαντήσεις. Πρώτον, η δική μας σφαίρα, εκεί που έχουμε αναλάβει κάποια δράση επιτόπου, ε, τοπικά σε τοπικό επίπεδο και το τι κάνει το προσωπικό μας εκεί και θεωρώ ότι αυτό ήταν ένα πρόβλημα σε πολλές αποστολές και κατά πάσα πιθανότητα εσείς ε, σε συνεργασία με εμά και αυτούς που κατευθύνουν τις αποστολές δεν μπορούμε παρά να απευθύνουμε μια έκκληση προς τις χώρες μέλη να παράσχουν τα στελέχη, να προβούν στη στελέχωση του προσωπικού ή είναι το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το οποίο έχει αξιοποιηθεί στις αποστολές αυτές. Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Άρα η ερώτηση έχει ως εξή. Ε, υπάρχει κάποιος μηχανισμός προκειμένου να μπορέσουν οι χώρες μέλη να είναι πιο προετοιμασμένες να παράσχουν το αναγκαίο προσωπικό. Ε, αυτή, γιατί αυτή τη σφαίρα μπορούμε εμείς άμεσα να την επηρεάσουμε. Από την άλλη πλευρά... Ε, τι είπαν οι δικοί μας άνθρωποι που βρίσκονται εκεί, τι σας είπαν σε σχέση με την ετοιμότητα, την ε, ε, κατανόηση εκ μέρους των αρχών του Μαλή και της Νιγηρίας ότι υπάρχει μια, όχι μόνο μια βούληση αλλά και μια ικανότητα να φτιάξουν τα πράγματα οι αμφιβολίες μας αμφιβολίες αφορούν την ε, βασική ε, ικανότητα και ίσως την ε, διάθεση να πράξουν αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους, να αυξηθεί η διοικητική τους ικανότητα, να πληρωθούν ε, οι θέσεις εκείνες για τις οποίες προβλέπονται αυτές οι δομές. Θα ήθελα να μάθω τι σας είπαν τα στελέχη, κατά πόσο υπάρχουν ανησυχίες αυτούς που είναι επιφορτισμένοι στις χώρες αυτές, κατά πόσο ε, συναισθάνονται την ανάγκη, την καταπήγουσα ανάγκη να κάνουν κάτι. Ή αλλιώς ε, ή, ή λένε απλώ, εντάξει κάντε ό,τι μπορείτε, ε, αν τα πράγματα πάνε καλά, έχει καλός, αυτά. Έχετε την αίσθηση ότι κάπως έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Στην αρχή είπατε βραδία πρόοδος. Γιατί όμως, αν υπήρχε πολιτική βούληση θα υποθέταμε ότι θα σημειωνόταν πιο ουσιαστική πρόοδος. Γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει αρκετό ζήλος από την άλλη πλευρά, δέσμευση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Μανόρτεν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ από ό,τι ξέρω καμία από αυτές τις αποστολές ε, δεν έχει υποστεί κανονικό έλεγχο και από την άποψη της οργάνωσης αλλά και από την άποψη την επιχειρησιακή. Βεβαίως ε, αυτοί οι οποίοι δέχονται αυτή τη στήριξη θέλουν τα μέσα και τα κονδύλια να φτάνουν μέχρι αυτούς. Οι βασικές αξίες, από ό,τι καταλαβαίνω από άποψη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι να παρουσιάζει όλα τα θετικά αυτών των αποστολών ε, με εντυπωσιακέ στατιστικές που ουσιαστικά εντυπωσιάζουν μόνο αυτούς που δεν γνωρίζουν Τελικά βλέπουμε όμως ότι αναλαμβάνουμε μία ευθύνη, ότι χρηματοδοτούνται με ευρωπαϊκά κονδύλια, ότι ενδεχομένως συμμετέχουν και άλλοι σύμμαχοι οι οποίοι νομίζουν ότι συμμετέχουν σε μια εξαιρετικά αποτελεσματική ε, αποστολή ε, στο Σαχέλ και βλέπουμε ότι τελικά είναι γαλλική αποστολή ότι τελικά πρόκειται για σχέδια CSDP τα οποία τελικά όμως ουσιαστικά δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς τι πάει που. Σήμερα στις Βρυξέλλες έχουμε την ψευδέστηση ότι πρόκειται για ευρωπαϊκές ε, αποστολές. Υπάρχει η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ αυτές τις μέρες και καταλαβαίνετε ότι εκεί είναι ξεκάθαρο ότι αν το ΝΑΤΟ δεν θέλει να εμπλακεί σε κάποιες περιοχές θα πρέπει κάποιος να καλύψει αυτό το κενό. Το γεγονός όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δημιουργήσει όλο αυτό το ε, σύστημα, ενδεχομένως θα πρέπει να το εξετάσουμε και να δούμε ποιος εξυπηρετεί συμφέροντα ποιου. Πριν ξαναδώσω στην κυρία Γιάκοψεν το λόγο, θα ήθελα να σας πω ότι διαβάζοντας αυτή την έκθεση βεβαίως δεν ήμουν εξαιρετικά ευτυχής, δεν ήταν πολύ ευχάριστο. Είναι η τρίτη συνάντηση που έχουμε για αυτό το θέμα, για τέτοιες αποστολές και πρέπει να σας πω ότι και με τον ε, κύριο Στίβενς, τον ε, πρέσβη, του ζήτησα την ε, δική του αν θέλετε, άποψη όσον αφορά αυτές τις αποστολές στην περιοχή της Σαχάρας, κοινέ αποστολές. Σκοπός μας είναι να υπάρξει μια περαιτέρω δέσμευση των ε, τοπικών κυβερνήσεων και δυνάμεων από τις χώρες τις οποίες λαμβάνουν χώρα αυτές οι αποστολές. Σίγουρα χρειάζεται πιο σοβαρή αξιολόγηση, μεγαλύτερη συμμετοχή από τις τοπικές κυβερνήσεις. Ποιος εκπροσωπεί την Επιτροπή, τι μπορείτε να μας πείτε. Καλημέρα σας, ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μας καλέσατε. Ήδη είχαμε αρκετές συζητήσεις με το ελεγκτικό συνέδριο. Ναι, όπως σας είπα είχαμε ήδη συζητήσεις με το ελεγκτικό συνέδριο κατά την προετοιμασία της έκθεσης αυτής. Όλες οι απαντήσεις μας, ε, οι απαντήσεις της Επιτροπής πώς βλέπουμε εμείς τα πράγματα και τις συστάσεις. Δεχόμαστε σε γενικές γραμμές τα συμπεράσματα και τις συστάσεις αυτής της έκθεσης. Θεωρούμε ότι είναι χρήσιμες, ήδη τις επεξεργαζόμαστε, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για δείκτες, καλύτερα συστήματα αρχαιοθέτησης, αξιολόγηση της προόδου, παρακολούθησης και εποπτείας. Συμφωνούμε με όλα αυτά, τα λαμβάνουμε υπόψη μας και είμαστε στην φάση της ενσωμάτωσης. Πιστεύω το ίδιο κάνει και η Επιτροπή. Δεν θέλω όμως να μιλήσω εξ ονόματος Επιτροπής. Η μεθοδολογία για τις μετρήσεις που χρησιμοποιήθηκε από το ελεγκτικό συνέδριο που οδήγησε εξάλλου και σε αυτόν τον τίτλο που μας φαίνεται λίγο αυστηρός, αντιστοιχεί στην σωστή κατά την άποψή μας μεθοδολογία για την αξιολόγηση τέτοιων ε, σχεδίων και προγραμμάτων. Χρησιμοποιείται και σε άλλες ε, περιπτώσεις. Απλώς, όσον αφορά ουσιαστικά μία τέτοια αποστολή ε, ασφάλειας στην περιοχή αυτή της Σαχάρας, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η διάρκεια, ο χρόνος που είναι πολύ μεγαλύτερος Χρειάζεται οπωσδήποτε και πολιτική βούληση και συμμετοχή των κρατών και των κυβερνήσεων επιτόπου. Η κατάσταση δεν είναι ίδια στην, στον Ήγυρα και στο Μαλί. Οι δυνάμεις ε, στο Νίγηρα είναι πολύ δεσμευμένες και πολύ αποφασισμένες όσον αφορά την τήρηση των συστάσεων και όσον αφορά την τήρηση ε, της τάξης. Έχουν μια αποστολή ασφάλειας. Στο Μαλί τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Με άλλες, αν θέλετε, δυνάμεις, την δύναμη μηνούσμα, επιτόπου κτλ. Και δεν είναι εύκολο να μετρηθεί η δράση και οι επιπτώσεις επιτόπου στο Μαλί. Παρ' όλα αυτά, αυτές οι δύο αποστολές έχουν ε, στηριχθεί και έχουν ε, επιβεβαιωθεί και συνεχιστεί από τις κυβερνήσεις επιτόπου, από τα συμμετέχοντα κράτη και νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η δράση τους καθώς και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γιάκοψεν για να απαντήσει στις ερωτήσεις και τα σχόλια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι ο κύριος Γκάλερ ρώτησε για ένα μηχανισμό προετοιμασίας των εμπλεκόμενων, του προσωπικού, των συμμετοχόντων σε αυτές τις αποστολές. Και βλέπουμε από την έκθεση των ελεγκτών ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει κίνητρο για πιο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Και η Επιτροπή και η Επιτροπή Εξωτερικής Δράσης σίγουρα θα πρέπει εδώ να επεκτείνουν τη χρονική περίοδο κατά την οποία το προσωπικό μένει επιτόπου. Πρέπει όμως να δούμε και τον ετήσιο προεπολογισμό γιατί σίγουρα με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αυξηθεί το κίνητρο, αν υπάρχει δηλαδή μια καλύτερη προοπτική χρονική μπορεί το προσωπικό να δεσμευτεί για περισσότερο χρόνο και να είναι και πιο αποτελεσματική η δράση τους επιτόπου. Τώρα, όσον αφορά τη διάθεση των ε, χωρών επιτόπου, την πολιτική τους βούληση για στήριξη, νομίζω ότι εδώ είναι πολιτικό το θέμα. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι τοπικές κυβερνήσεις δέχονται τις απαραίτητες αλλαγές ε, στην νομοθεσία τους, παραδείγματος χάρη. Η επιβολή συγκεκριμένων ε, συνθήκων, η στήριξη από μέρους ε, των κρατών αυτών σε μια αποστολή που σαφώς θα πρέπει να στηριχθεί από τις τοπικές κυβερνήσεις υπό προϋποθέσεις. Θα πρέπει λοιπόν να θέσουμε σαφείς προϋποθέσεις και όρους στην βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη στήριξή της. Κύριε Βαν Όρτανελ, μιλάτε για ψευδέστηση, μιλάτε για ε, την εικόνα που δίνεται. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου εμείς ελέγχουμε ουσιαστικά τα αποτελέσματα, την αποτελεσματικότητα. Φυσικά και όλοι θα θέλαμε καλύτερα συμπεράσματα, πιο θετικά για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Για τη μεθοδολογία. Εγώ εκπλήσωμαι λίγο από αυτά που είπε η εκπρόσωπος ε, της υπηρεσιτητής εξωτερικής δράσης. Γιατί να υπάρχει ειδική μέθοδος μέτρησης όταν πρόκειται για την Επιτροπή. Υπάρχει στρατηγική, αν θέλετε, διάσταση σε αυτές τις συγκεκριμένες αποστολές που δεν υπάρχει αλλού. Πιστεύω ότι κάτι εδώ δεν πάει καλά με τη δική σας μεθοδολογία, γιατί πραγματικά σχεδιάζετε προγράμματα τα οποία περιμένουμε να έχουν κάποιο αποτέλεσμα και σε αυτή την περίπτωση τα στηρίζουμε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Γιάκοψεν. Θέλει κάποιος άλλος να πάρει τον λόγο. Όχι. Α, ο κύριος Γκάλερ. Ναι. Στην ετήσια έκθεση ήδη είχαμε επικρίνει όλες τις αποστολές λέγοντας ότι μόνο το 75% των θέσεων είναι καλυμμένες από προσωπικό. Τελικά λοιπόν βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη αποφασίζουν να συμμετάσχουν σε τέτοιες αποστολές και κατόπιν δεν καλύπτουν τις θέσεις με το απαραίτητο προσωπικό. Πρέπει να βελτιωθούμε σε αυτό το τομέα. Όλοι εμείς τα κράτη-μέλη. Και να μπορούμε να καλύψουμε με προσωπικό όπως υποσχόμαστε. Και βεβαίως να είμαστε και πιο αποτελεσματικοί επιτόπου. έτσι ώστε αυτοί που πρέπει να αναλάβουν αυτές τις αποστολές να το κάνουν με αποτελεσματικότητα θέλω να συμμετέχουν και τα κράτη να αναλάβουν αν θέλετε την καλύτερη διαχείριση και διοίκηση των ε, κρατών τους, των υπηρεσιών τους και να δώσουν μια καλύτερη εικόνα στους πολίτες τους. Εμείς βεβαίως πρέπει να λειτουργήσουμε με κίνητρα, με επιβράβευση και με αυστηρότητα. Και όχι να αφήνουμε τα πράγματα να εξελιχθούν και κατόπιν να λέμε ξαφνιάζουμε γιατί τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που θα θέλαμε. Αυτό δεν είναι λύση. Η αξιολόγηση και οι μετρήσεις, αν θέλετε, δεν πρέπει να γίνονται μόνο στο χαρτί και διοικητικά, αλλά επιτόπου αν το αποτέλεσμα είναι θετικό για τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ έχω θίξει το θέμα αυτό, του πώς θα καλυφθούν οι θέσεις με το αρμόδιο προσωπικό. Το συζήτησα και με τον ε, πρέσβη, τον κύριο Στίβενς. Συζήτησα και με την γραμματεία για το θέμα της παρακολούθησης όλων των αποστολών. Γιατί σε γενικές γραμμές αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι όταν είμαστε παρόντες σε κάποιες τέτοιες αποστολές, αποστολές της ε, Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας, και στο Νίγηρα και στο Μαλί και στην Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής. Όπου είμαστε λοιπόν παρόντες, διαπιστώνουμε προβλήματα και ατασταλίες. Και το πρώτο τμήμα της παρουσίασης της κυρίας Γιάκοψεν μας δείχνει ξεκάθαρα ότι σε σύγκριση με άλλες αποστολές, οι αποστολές Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζονται με πολύ καλύτερο τρόπο από τις ε, τοπικές αρχές, από τα κράτη. Παρόλα αυτά, πρέπει να έχουμε καλύτερη αξιολόγηση Είμαστε ίσως το καλύτερο σχήμα για να ασκήσουμε πίεση επιτόπου στις αρχές των κρατών αυτών και ως ε, Επιτροπή Εξωτερικής Δράσης αλλά και ως Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να παρουσιάσουμε το έργο μας αλλά δεν είναι δικός μας ρόλος να κάνουμε τον έλεγχο εις βάθος. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια. και ευχαριστούμε πολύ και την Επιτροπή και τους εκπροσώπους. Ελπίζουμε να έχουμε και άλλες επαφές μαζί σας. Okay, I have to announce break until uh, 3.30.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 Yeah.

πρωτάθλημα.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

Colleagues, Κυρίες και κύριοι, ας ξαναξεκινήσουμε. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι οι αποστολές ε, ΚΕΠΑ και επιχειρήσεις για θέματα σταθεροποίησης στο κέρας της Αφρικής. Με χαρά καλωσορίζω τα μέλη του πάνελ. πλήρχος Ντανιέλε Μαρτινούτσι. Εκπροσωπεί το Ιταλικό Ναυτικό. Μάλλον την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Εξεβονίμων. Η κυρία Σεάννα Λάκ που ε, εκπροσωπεί το CCP. Η προηγούμενη Ολομέλεια ασχολήθηκε με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα κατεπήγοντα, την κατεπήγουσα κατάσταση, την κατάσταση ανάγκης στη Σομαλία, ετέθηκε το θέμα της ασφαλείας στη χώρα. Συχνά στη θητεία έχουμε συζητήσει τα θέματα ασφαλείας στο κέρας της Αφρικής. Επισκεφθήκαμε το αρχηγείο της ναυτικής αποστολής Αταλάντη στο, στη Βρετανία. Ξέραμε ότι εν ώψη του Brexit χρειάζεται μία ε, ανακατάταξη της οργάνωσης των αποστολών και το αρχηγείο θα μετακινηθεί από το Λονδίνο και θα πάει ίσως θα πάει σε Γαλλία μάλλον στη Ισπανία βασικά και ίσως κάποιο τμήμα και στη Γαλλία θα ληφθούν αργότερα οι τελικές αποφάσεις να δώσω αμέσως το λόγο στον ε, Πιέρχο Μαρτινούτσι να παρουσιάσει τις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι ο Ντανιέλε Μαρτινούτσι, πλήρχος Ιταλικού Ναυτικού. Και είμαι, είμαι αποσπασμένος ε, εμπειρογνώμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο στρατιωτικές δραστηριότητες ΚΕΠΑ είναι στο Λαβάν στο κέντρο της Αφρικής μια εκτελεστική αποστολή, η επιχείρηση Αταλάντη και μια μη εκτελεστική εκπαιδευτική αποστολή. UTM Σομαλία. Και οι δύο αποστολές έχουν εντολή που εκπνέει την 31η Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους και σύμφωνα με την στατηγική έκθεση που ενέκριναν τα κράτη-μέλη και οι δύο αποστολές έχουν τύχει επέκτασης της εντολής για μία ακόμα διετία. Όσον αφορά την εκπαιδευτική αποστολή στη Σομάλια, στόχος είναι το να συμβάλλουμε την αύξηση δυνατοτήτων στη Σομαλία, στον τομέα της ασφάλειας, στον αμυντικό τομέα. Γενικός στόχος να ενισχυθεί όλη η δομή του Σομαλικού Υπουργείου Αμήνης και του Γενικού Αρχηγείου των Ενόπλων Δυνάμεων και έτσι να μπορέσουν οι Σομαλοί να εκπαιδεύουν ε, τις ένοπλες δυνάμεις Σομαλίας. Άλλο στόχος της αποστολής. Να αυξηθεί η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κέρας Αφρικής. Στο Μογκαντήσο ενεργοποιείται η αποστολή. Αλλά υπάρχει και έμεση διάδραση ε, με άλλες αποστολές ε, και προγράμματα της ΚΕΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί. Η αποστολή στηρίζεται από 8 κράτη-μέλη και μία τρίτη χώρα τη Σερβία έχουμε 170 ανθρώπους που εργάζονται στα πλαίσια αυτά στο Μαγκαντήσου είναι εκπαιδευτική αποστολή που σας είπα σχεδιάζεται και εφαρμόζεται ε, στις Βρυξέλλες, στα πλαίσια του στατιωτικού σχεδιασμού. Γίνεται αναθεώρηση της αποστολής τώρα Εξετάζουμε τα έγγραφα σχεδιασμού για να υποβληθούν προς έγκριση τα κράτη-μέλη και μετά να υποβληθούν στο Συμβούλιο για να έχουμε πλήρη έγκριση της επέκτασης της εντολής από 1η Πρώτου 2019 μέχρι 31η Δεκεμβρίου του 2020. Η επόμενη θητεία θα προσαρμοστεί κάπως για να αλλάξει κάπως η πορεία της αποστολής της εκπαίδευσης ούτω ώστε να αναθέσουμε περισσότερα καθήκοντα στους ομαλούς εκπαιδευτές μέχρι να αναλάβουν ποιος αυτήν την αποστολή και η βασική αποστολή θα μετατραπεί σε συμβουλευτική. Θα βοηθούμε το Υπουργείο Αμήνας που τελικά θα ηγούνται του Υπουργείου Αμήνης ε, πολίτες, πολιτικοί και θέλουμε να διευκολύνουμε το σχεδιασμό ε, της αλλαγής αυτής για να γίνει όλη η διαδικασία από τον Σομαλικό στρατό. Έχουμε την εκτελεστική μετά αποστολή, την ε, επιχείρηση Αταλάντα. Η, Πολιτική και Στρατιωτική Επιτροπή δέχτηκε παράταση για μία διετία από 1η του 2019 μέχρι 31 Δωδεκάτου του 2020. Εξετάζουμε όλα τα έγγραφα σχεδιασμού για αυτή την επιχείρηση και θα παραλάβουμε το νέο σχέδιο, δεν άλλαξε η εντολή. Αφορά την προστασία παράδοσης προμηθειών από το παγκόσμιο σύστημα τροφοδοσίας, παροχής τροφίμων στο Μαγκαντήσου και να αποτρέψουμε τις επιθέσεις των πειρατών. Και Είμαστε σε επιφυλακή για να δραστηριοποιηθούμε τυχόν υπάρξει ε, δραστηριοποίηση των ε, πειρατών. 20 κράτη-μέλη συμμετέχουν σε αυτή την αποστολή και τρεις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσης, Μαυροβούνιο, Σερβία και πρόσφατα συμμετέχει και η Δημοκρατία της Κορέας. Δύο πλοία και ένα αεροσκάφος ε, θαλασσίων ε, αποστολών μακράς εμβελίας συμμετέχουν και όπως είπε η κυρία Πρόεδρος λόγω της απόσυσης ενός κράτους μέλους από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα λάβει χώρα τον επόμενο Μάρτιο που έχει, που έχει ένα κατέχει ένα από τα αρχηγεία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως έχουν προσφορές από Γαλλία και Ισπανία για να μπορέσουν να ηγηθούν ε, των μελλοντικών ε, επιχειρήσεων. Αυτή είναι η κατάσταση. Περιμένουμε λοιπόν τα διάφορα έγγραφα που θα αφορούν το σχεδιασμό. Ε, Πλήρχε, μπορείτε να μας πείτε περισσότερα πράγματα για την κατάσταση γενικότερα για την ασφάλεια. Το περιβάλλον, σε την ασφάλεια και ποιο είναι το περιβάλλον στο οποίο κινούνται οι δύο επιχειρήσεις. Ναι, κυρία μου. Για την ασφάλεια. Οι δύο στατητικές επιχειρήσεις αυτές επιδούν η μία επί της άλλης. Από τη μία έχουμε την εκπαίδευση, γίνεται σε χερσαίο στην, στην Ξηρά, στην περιοχή του Μογκαντήσου. Εξετάζουμε θέματα που αφορούν το πολιτικό πεδίο, το Υπουργείο Άμυνας και με το στρατηγείο και με το στατικό προσωπικό. Μετά έχουμε την επιχείρηση Αταλάντα, που είναι θαλάσσια, που έχει όμως θετικό αντίκτυπο όσον αφορά τις επιχείρησης και οι δύο θετικές επιχειρήσεις αλληλοενισχύονται. Η εκπαιδευτική επιχείρηση Σομαλία αντι... αντιμετωπίζει περισσότερα προβλήματα ασφαλείας. Διότι το περιβάλλον είναι εύθραυστο όσον αφορά την ασφάλεια στη Σομαλία. Δεν έχει γίνει πλήρης αξιολόγησης από τους Σομαλούς. Τι εννοώ η συνταγματική δομή, η νέα συνταγματική δομή που υπάρχει. Σε επίπεδο ομοσπονδιακής κυβέρνησης και ομοσπόνδων κρατών χρήζει συμφωνίας. Δεν έχει ξεβρεθεί ακόμα συμφωνία. Η διεθνής κοινότητα έχει καταβάλει πολλές προσπάθειες για να επιτευχθεί συμφωνία. Σε αυτή τη φάση πιστεύουμε ότι υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία καταρχάς σε πολιτικό επίπεδο και μετά αυτό έχει και αντίκτυπο στην ασφάλεια. Η ασφάλεια Η κατάσταση φορά την ασφάλεια είναι περίπλοκη. Πολλοί θέλουν να συμβάλλουν στην αποκατάσταση της σταθερότητας στην περιοχή. Και όλοι οι διεθνείς φορείς προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο συντονισμού μεταξύ τους και έτσι να συμβάλλουν ενεργά στη γενική προσπάθεια. Γι' αυτό το σκοπό λειτουργεί η γενική διευθέτηση για την ασφαλεία που συμφωνήθηκε το 2017 από τη Διεθνή Κοινότητα στο Λονδίνο, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στρατιωτικός κλάδος συνεργάζεται με τη ΣΥΠΑ. Θέλουμε να αυξηθεί η ασφάλεια για τον Εθνικό Στρατό της Σομαλίας. Έχουμε και επίση για το κάτω δικαίου την 2 Τσάρλι και μια άλλη υποστολή που αφορά τι ένοπλε δυνάμει. Αυτή είναι η γενική εικόνα ε, και έχουμε την πεποίθηση ότι έχουμε βελτίωση. Ευχαριστώ, Πλήρχε. Κυρία Λάκας, ε, μας μιλήσει τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Θα σας κάνω μια παρουσίαση για την Γιούκο από τη Σομαλία και το ρόλο της όσον αφορά την ε, δημιουργία της ασφάλειας ε, σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο στη Σομαλία. Θαλάσσια ναυτική ασφάλεια για τις αρχές της ε, Σομαλίας, τα λιμάνια της Σομαλίας ξεκινήσαμε το 2002, αν θυμάστε, ξεκίνησε με την πρώτη αποστολή για τη δημιουργία δυνάμεων θαλάσσιων στην περιοχή και στον Ινδικό ωκεανό, στο κέρας Αφρικής. Επρόκειτο για μια αποστολή η οποία δεν ήταν πάρα πολύ ικανοποιητική. Υπήρξαν κράτη-μέλη τα οποία ζήτησαν τότε να αναδιαρθρωθεί η όλη αποστολή, μετονομάστηκε σε UCAP Σομάλια και α, στόχευε την δημιουργία μιας δύναμης μόνο για τη Σομαλία και όχι για όλη την περιοχή. Στηρίζουμε τις αρχές ε, της Σομαλίας και θα σας εξηγήσω ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους είναι απαραίτητη η ε, ασφάλεια στην θάλασσα για την χώρα αυτή τη Σομαλία. Έχει μια πάρα πολύ σημαντική ακτογραμμή, τη μεγαλύτερη στην περιοχή αυτή της Αφρικής. Έχει δηλαδή πολύ μεγάλα θαλάσσια σύνορα. Είναι λοιπόν προϋπόθεση να εγγυηθεί κανείς ε, την ασφάλεια στη θάλασσα και την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Η Σομαλία δεν έχει αρκετές δυνάμεις θαλάσσιες αυτή τη ε, στιγμή έτσι ώστε να περιορίσει όλες ε, τις εγκληματικές ε, δραστηριότητες στην περιοχή αυτή και στις ακτές της. Η ίδια η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας παραδέχεται λαθρεμπόριο, πειρατή τικές ε, αποστολές, δραστηριότητες, επιχειρήσεις εγκληματικές στην περιοχή και στα χωρικά της ίδατα. Ε, υπάρχει λοιπόν ασφάλεια, συγγνώμη, υπάρχει έλλειψη ασφάλειας στην περιοχή, κάτι το οποίο ξεπερνάει τις δυνατότητες ε, της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας. Η οικονομική σημασία των λιμανιών σε καμία περίπτωση δεν πρέπει εδώ να υποτιμηθεί. Είναι πολύ σημαντικά τα έσοδα και για την Σομαλία και όσον αφορά τις αλλιευτικές άδειες και την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κάτι το οποίο θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και για τις επόμενες γενιές. Η ναυτική ασφάλεια λοιπόν, η θαλάσσια ασφάλεια, η λεγόμενη γαλάζια οικονομία είναι απαραίτητη και μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη της οικονομίας της Σομαλίας. Εξού και ξεκίνησε η ενίσχυση της επιχείρησης UCAP Σομαλία. Όπως είπε ο πλοίαρχος, τα τελευταία δύο χρόνια έχει προοδεύσει, έχει βελτιωθεί η κατάσταση στην Σομαλία με τη δημιουργία δομών και με μια ανασφάλεια η οποία δυστυχώς δεν έχει εξαλειφθεί και επηρεάζει την καθημερινή ζωή των πολιτών της Σομαλίας. Για γεωπολιτικούς ε, λόγους, για έλλειψη δημοσιονομικής σταθερότητας, η κατάσταση στη Σομαλία συνεχίζει από οικονομικής πολιτικής ε, απόψεως να παραμένει προβληματική. Έλλειψη πόρων και παράνομες ε, δραστηριότητες και ανάπτυξη είναι προκλήσεις οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Όσον αφορά την ασφάλεια που είναι καθοριστική όπως και στο παρελθόν, η οικονομική δραστηριότητα, η οικονομική ανάπτυξη, ιδιαίτερα στο, στην θάλασσα αλλά και στις ακτές, θα πρέπει να διασφαλιστούν. Η αποστολή Γιου Καψομάλια έχει σαν σκοπό να βοηθήσει την δημιουργία δομών και δυνάμεων σε αυτήν την δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στο, στις κρατικές δομές της Σομαλίας. Πρώτος μας στόχος είναι η στήριξη καλύτερης ε, διακυβέρνησης αρχών λιμενικών ε, στις ακτές αλλά και θαλάσσιας δύναμης. Δεύτερον, ενίσχυση των ε, δυνάμεων επιβολής του νόμου και ενίσχυση της επιχειρησιακής δύναμης στο ναυτικό και θαλάσσιο τομέα. Όσον αφορά τη διακυβέρνηση, όσον αφορά τη δημιουργία δομών και δυνάμεων για την επιβολή του νόμου, στην συνδιάσκεψη του Λονδίνου το Μάιο του 2017 ήταν ε, η πρώτη πολύ σημαντική απόφαση για την ε, Συμφωνία Ανάπτυξης και Στήριξης Δυνάμεων Ναυτικών ε, στη Σομαλία. Ουσιαστικά αυτό αποτέλεσε και τη βάση για την UCAP Σομάλια να ενισχύσει την παρουσία της, ε, τη δομές της, μετά από αυτές τις πολιτικές αποφάσεις, οι οποίες αρχικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ληφθούν. Οι δυνατότητες διακυβέρνησης ε, της ε, Σομαλίας των ε, θαλάσσιων ακτοπλοϊκών δομών είναι ακόμα σε αμβριακό στάδιο. Οι αποφάσεις που ελήφθηκαν στη συνδιάσκεψη του Λονδίνου και η ειδική ενίσχυση των δομών σίγουρα θα πρέπει να συνεχιστούν και να μην παραμείνουμε στις πρώτες αυτές αποφάσεις που δημιουργήσαν μια κινητικότητα. Είναι σημαντικό να συνεχίσει η αποστολή UCAP επιτόπου να στηρίζει με παροχή συμβουλών, με ενίσχυση δομών, με δημιουργία δυνάμεων και με την στήριξη διαδικασιών λήψης αποφάσεων η δημιουργία νέων δομών, θαλάσσιων, το νομικό πλαίσιο στο οποίο θα μπορέσουν να λειτουργήσουν οι θεσμοί αυτοί. Υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο στην ε, Σομαλία, το οποίο όμως είναι απαρχαιωμένο, παρουσιάζει σημαντικές αδυναμίες και είναι και ανεπαρκές. Υπάρχουν ε, συγκεκριμένες προτάσεις νομοθεσίας που προετοιμάζονται και αφορούν ε, τις θαλάσσιες ε, δομές. Βεβαίως χρειάζεται πολιτική βούληση. Η δράση της αποστολής σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τις αποφάσεις που θα ληφθούν επί από τις ε, αρχές της Σομαλίας όσον αφορά τις επιχειρησιακές δομές για την ε, ναυτική και θαλάσσια ασφάλεια. Ξεκινούμε από μία προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω, στήριξη δηλαδή των υπαρχόντων δομών και δημιουργία επιπλέον δυνατοτήτων. Μέχρι τώρα η αποστολή έχει στηρίξει όλες τις δομές, ε, τους οργανισμούς και τους φορείς που υπάρχουν και λειτουργούν ε, στο Μογκαντήσιο με προγράμματα που στηρίζονται ήδη για τη δημιουργία νέων θαλάσσιων δομών, ενίσχυση των υπαρχουσών δομών, Μπορούμε να πούμε επίσης ότι από τότε που το 2015 η UCAP Σομάλια ενισχύθηκε και μετονομάστηκε, έχει στηριχθεί από περισσότερα κράτη-μέλη, έχει ενισχυθεί και σιγά σιγά η αποστολή αυτή επανδρώνεται με το απαραίτητο προσωπικό έτσι ώστε να μπορέσει να είναι αποτελεσματική, να καλύψει όλο το εύρος των ε, διαφορετικών πτυχών με ένα γραφείο στο Λονδίνο και ένα επιτόπου. Αυτό χρησιμοποιείται με ένα επιτυχή τρόπο μέχρι τώρα, με έναν ρόλο μεσολάβησης και διευκόλυνσης. Για το μέλλον, τους επόμενους μήνες, χρειάζεται καλύτερη συνεργασία, κοινό σχεδιασμός με την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με τα εργαλεία επιτόπου για να επιτευχθεί περισσότερη αποτελεσματικότητα και επιτυχία. Χρειάζεται όμως και πολιτική στήριξη από την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιτόπου καθώς και συνεργασία με όλους τους συναδέλφους επιτόπου. Θα συνεχίσουμε τη στήριξη όλων των δομών για περισσότερη ασφάλεια στις θάλασσες και στις ακτές της Σομαλίας και την στήριξή μας για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Είναι σημαντικό να μεταφερθεί η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνδυασμό με τις ναυτικές δυνάμεις, με τις δυνάμεις που δρούν στις ακτές της Ομαλίας, είναι καθοριστικό για την επιτυχία της UCAP να παραμείνει σε στενή επαφή με την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και με την αρχιτεκτονική για την ασφάλεια όπως αποφασίστηκε στο Λονδίνο. Ευχαριστούμε πολύ. Ασφαλώς πάντοτε υπάρχει μια διασύνδεση μεταξύ ε, ασφάλειας και διαφόρων ε, δραστηριοτήτων σταθεροποίησης και αναπτυξιακής βοήθειας. Ε, και έχουμε ένα εκπρόσωπο εδώ της ΔΕΦΚΟ. Ίσως θα ξεκινήσουμε με τη δική του παρέμβαση. τη δική της μάλλον. Είναι εκτός μικροφώνου. Αισθάνεστε ήδη κάποιες ε, θετικές ε, επιπτώσεις όσον αφορά τις ε, εξελίξεις στην Αιθιοπία και την Ερυθρέα και τη σχέση μεταξύ Αιθιοπίας και Ερυθρέας. Ε, συγγνώμη, υπήρξε μια παρανόηση. Νόμιζα ότι ήταν ο εκπρόσωπο της ε, γενική διεύθυνση. Λάθος, ο κύριος Γκάλερ. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Όπως είπατε, από τη μία πλευρά υπάρχει αυτό το δυναμικό με την μακρά ακτογραμμή, την αλία κλπ. Και αν η χώρα ήταν σε θέση να διαχειριστεί την ε, ζώνη της, ε, ε, των 200 μιλίων και να μπορούσαν οι αλλοίς να διοδοθούν και να ασκήσουν κανονικά τις δραστηριότητές τους, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Θα μπορούσατε να ποσοτικοποιήσετε, να μας πείτε με αριθμούς τι γίνεται με την ακτοφυλακή, την θαλάσσια αστυνομία, ε, ποιο κομμάτι της ακτογραμμής αυτή τη στιγμή είναι στη θέση να ελέγξουν. Γιατί βορειοδυτικά έχουμε de facto το Somaliland, το οποίο είναι τμήμα του ημίσεως της ε, ακτογραμμής είναι αυτή η περιοχή μια περιοχή όπου οι de facto αρχές εκεί του Σομάλιλαντ ασκούν τα καθήκοντά της υπό τη έννοια ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν πλέον πειρατές που να προέρχονται από εκεί και ενδεχομένως θα υπήρχε δυνατότητα να δοθούν αλλιευτικές άδειε στην περιοχή αυτή γιατί πράγματι υπάρχει μια έδρα τη κυβέρνησης εκεί γιατί αυτό μας απασχολεί και συνολικά για πόσα άτομα μιλάμε όταν μιλάμε για κατάρριση του προσωπικού της εκτοφυλακής ή της αστυνομία, αλλά αστυνομία. Και ποιες είναι οι αποδοχές τους. Μπορεί η κυβέρνηση να τους αμείβει κανονικά. Ας ελπίσουμε ότι αυτό δεν είναι θέμα και θα ακούσουμε ότι έχει δηληθεί. Αυτά. Είπατε, αναφερθήκατε στους πειρατές και στις τρομοκρατικές ομάδες, στην Αλσαμπάμπ και λοιπά. Δεν έχουμε τις δικές μας δορυφορικές ε, ικανότητες να κάνουμε αυτή την ανείχνευση. Η UCAP, η Αταλάντα θα μπορούσε να τις αξιοποιήσει προκειμένου να ανοιχνεύσει τους κινδύνους όσον αφορά τις δικές μας αναπτυξιακές Κυρία Γκόμες, ε, θέλετε να προσθέσετε εσείς τη δική σας ερώτηση, αλλιώς θα υποβάλω εγώ μια ερώτηση και στη συνέχεια θα απαντήσουν οι ομιλητές και ο εκπρόσωπος της ΔΕΦΚΟ. Θα θέλετε εσείς να πάρετε το λόγο. Νομίζω ότι εξελίξει σε αυτή την περιοχή του κόσμου θα μπορούσα να είναι πολύ σημαντικές για τη Σομαλία και για την ασφάλεια στα ύδατα της Σομαλίας και για τον Νότιο Σουδάν επίσης, λόγω του ρόλου που διαδραματίζει η Αιθιοπία εκεί. Αναμένεται και κάποιες θετικές εξελίξεις ένα από τα δικά μου ερωτήματα μοιάζει με την ερώτηση της Γκόμες. Είναι το εξή. Θα ήθελα να ρωτήσω, ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, αποχώρηση της αποστολής Αμισόμ από τη Σομαλία. Ποια είναι, ποιο είναι το προγραμματισμένο modus operandi δέσμευση σε χώρες όπως είναι η Αιθιοπία η Κένια όχι μόνο σε άλλες περιοχές, αλλά και όσον αφορά τις προσπάθειες σταθεροποίησης στην Αιθιοπία. Γιατί και εκεί ε, ήταν παρουσία μισό. Ποιο είναι λοιπόν το πραγματισμένο, πραγματιστής τρόπος λειτουργίας των ειρηνευτικών και προσπαθειών και των προσπαθειών σταθεροποίησης της περιοχής. Ο πρόεδρος Μοχάμετ δήλωσε ότι έχει εξαλειφθεί, έχει αποδιαρθωθεί η Σαμπάμπ. Αλλά πρόσφατα πληροφορθήκαμε για κάποιες επιθέσεις τρομοκρατικής φύσεως, ευρείας κλίμακας όπως το Μογκαντήσου ή και άλλες ε, μικρότερες επιθέσεις. Ποιο είναι το πρόγραμμα το οποίο έχετε κατά νου προκειμένου να αναλάβετε ενεργό δράση στην πλατύτερη, στην ευρύτερη περιοχή. Παρακαλώ. Κάπτεν Μαρτίνο Τσίν, η κυρία Λάκ και στη συνέχεια η εκπρόσωπος της ΔΕΦΚΟ. Με συγχωρείτε που δεν γνωρίζω τα ονόματα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα αποφεληθώ. Από Θα απαντήσω τελευταία ερώτηση σχέση με τη δέσμευση που έχουμε στην μεταβατική περίοδο και τη μετατόπιση της ευθύνης στους ίδιους τους Ομαλούς. Την ανάθεση ευθύνη ομαλού. Υπήρξαν εδώ κάποιες εξελίξεις και έχει υπάρξει και μία συμφωνία η οποία οδήγησε σε ένα πρόγραμμα μετάβασης το οποίο αποτελεί ένα είδος μοντέλου και σχεδιάζοντας ακριβώς αυτό το πρόγραμμα μετάβασης λάβαμε υπόψη την ομάδα η οποία ε, είχε επιφορτιστεί ακριβώς με το σχεδιασμό αυτού του μοντέλου μετάβασης. Βεβαίως εδώ συμμετείχε και η διεθνή κοινότητα και η δική μας αποστολή ε, υποστήριζε την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήταν η ΙΠΑ, η Τουρκία και άλλοι συμμετείχαν προκειμένου να εξολογήσουν ποιο θα ήταν το δικό τους μερίδιο ευθύνης προκειμένου να γίνει ακριβώς αυτή η μετάβαση και να μπορέσουν οι σομαλικές μονάδες να αναλάβουν ευθύνη. Επειδή αναφερθήκαμε σε αριθμούς προκειμένου να αντικατασταθούν οι ομάδες της Νοτιοαφρικής ε, και να μπορέσει το, ο στρατός της Σομαλίας να αναλάβει. Γιατί κάποιες τοπικές ε, δυνάμεις μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο και υπάρχει μια γενική συμφωνία για όλους όσοι συμμετέχουν σε τη διαδικασία μετάβασης Έχουν, είχαν προσκληθεί όλοι, την έδρα είχε ο πρόεδρος ο κ. Μάντζο. Όσον αφορά την Αλσαμπάμπ, πράγματι είναι παρούσα στην περιοχή και πάντοτε προσπαθεί προκειμένου όχι μόνο να αισθητή την παρουσία της, αλλά και να αναγνωριστεί όχι μόνο από τους Σομαλούς, αλλά και από τη διεθνή κοινότητα. είναι δύσκολο να αξιολογήσουμε την ε, παρουσία της Al-Shabaab. Ε, γιατί υπάρχουν ε, δυσκολίες όσον αφορά τις πληροφορίες και την αποστολή κατάρτισης και την Αταλάντα. Η αποστολή κατάρτισης μετέβη εκεί κατόπιν πρόσκλησης κυβέρνησης αλλά δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες. Στη φάση αυτή η ανάπτυξη του, εκπόνηση του νέου σχεδίου για την Αταλάντα είναι να υπάρξει στοχεύει προς την ε, παροχή περισσότερων ε, πληροφοριών και διεξάγεται μια εκστρατεία σε σχέση ακριβώς με την ανταλλαγή ε, πληροφοριών. προκειμένου να χαρτογραφηθεί συνολικά το τοπίο στη Σομαλία και να αποθηθεί η Αλσαμπάμπ. Όσον αφορά το άλλο ερώτημα, νομίζω δεν είμαι αρμόδιος όσον αφορά την ανάπτυξη. Αυτό αφορά την EUCAP. Mm. Η κυρία Λακ. Φοβούμαι ότι και εγώ δεν είμαι πιο αρμόδια από εσά όσον αφορά τη στρατηγική ανάπτυξη στην περιοχή. Θα έπρεπε να απευθύνετε την ερώτηση σε πιο αρμόδιους. Όσον αφορά το κατά πόσο μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε την ε, ικανότητα διαχείρισης της ακτογραμμής, είναι δύσκολο να απαντηθεί αυτή η ερώτηση. Βεβαίως ε, θα πρέπει να πούμε ότι είναι ισχνή. Στο Μογκαντήσου είναι πολύ περιορισμένη αυτή η ικανότητα. Στο Σομάλιλαν τα πράγματα είναι καλύτερα. όπου υπάρχει το MPF. Είναι μια αστυνομική δύναμη που έχει το μεγαλύτερο δυναμικό, την μεγαλύτερη ικανότητα στην ε, περιοχή αυτή και είναι σε θέση να περιπολούν και να ελέγχουν τα χωρικά του ύδατα. Τώρα, για πόσα άτομα μιλάμε. Όταν αφορά την παρακολούθηση της ε, ακτοφυλακής, είναι δύσκολο να το πούμε γιατί η ακτοφυλακή δεν έχει σταθεί ακόμα και το MPO υπάρχει μόνο σε ορισμένα ομοσπονδιακά κρατήδια. Δεν πρόκειται για τεράστια νούμερα, ίσως ε, κάποιες δουζίνες, το πολύ 100, αλλά όχι πάνω από 100. Όσον αφορά την ασφάλεια και το πώς ε, θα μπορούσε κανείς ε, να ανοιχνεύσει τις κινήσεις των πειρατών. Νομίζω δεν είμαι αρμόδια να απαντήσω. Όσον, απα... όσον αφορά τη μετάβαση των... τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων της Αμισόμ στους Σομαλούς, δεν υπάρχει καθόλου ικανότητα ε, θαλάσσιας ε, διαχείρισης και θα πρέπει να οικοδομηθεί η ικανότητα αυτή εκ του μηδενός. Θα ήθελα να ζητήσω από την ε, εκπρόσωπο της ΔΕΦΚΟ να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν αρκετά θέματα. ακούσαμε ενδιαφέρουσες πληροφορίες που θα είναι χρήσιμες για τη συζήτηση. Δεν είμαι σίγουρη αν αναφέρθηκε από το Κοινοβούλιο, αλλά την προσεχή εβδομάδα έχουμε το φόρουμ εταιρική σχέση με τη Σομαλία, που είναι η άμεση παρακολούθηση συνδιάσκεψης του Λονδίνου, που ανέφεραν ε, οι βουλευτές και στη συνάντηση αυτή που ελπίζω θα είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο θα εξετάσουμε τρεις ε, πτυχές του μέλλοντος της Σομαλίας το πολιτικό μέλλον, την ασφάλεια που θα συμπεριλαμβάνει συζητήσεις σε σχέση με την αμισόμ και την μελλοντική χρηματοδότηση στο επίπεδο της ασφάλειας και την οικονομική ανάπτυξη. Όσον αφορά την πλευρά της οικονομικής ανάπτυξης, η Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ ήδη παρέχει σημαντική συνδρομή προς τη Σομαλία και πρόσφατα συμφώνησε 100 εκατομμύρια επιπρόσθετο προπολογισμό για την υποστήριξη του προπολογισμού και 83 εκατομμύρια για την σταθεροποίηση της κοινωνίας των πολιτών. Όσον αφορά τα προγράμματα θαλάσσιας ασφάλειας τα οποία ήδη αναφέρθηκαν, θα γίνει στο φόρουμ την επόμενη εβδομάδα, θα γίνουν κάποιες συζητήσεις με την Ιθιοπία και την Ερυθρέα και η εξέλιξη στη σχέση μεταξύ Ερυθρέας και Αιθιοπίας είναι εξαιρετικά ευπρόσδεκτη και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτή τη διαδικασία. Αναφέρεται ότι ενδεχομένως η Ερυθρέα θα μπορούσε να επιστρέψει στην ΙΓΚΑΝΤ. Ε, θα υπάρξουν πολλές αλλαγές γιατί με τον τρόπο που συμμετείχε η Αιθιοπία στο παρελθόν στην ΙΓΚΑΝΤ εάν αποφασίσουν να ε, παραδώσουν την ε, Προεδρία, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην έναρξη ενό περιφερειακού διαλόγου. Και αν αυτό συμβαίνει, θα ασχοληθούμε πολύ στενά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και την επικεφαλή κυρία Μογκαρίνη, η οποία είχε συζητήσει την περιοχή αυτή και η οποία προγραμματίζει μια άλλη συνάντηση τον Οκτώβριο. Την είχε ήδη προγραμματίσει πριν από τι πρόσφατε εξελίξει εντό τη Αιθιοπία. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα θα εστιαστούμε στη Σομαλία. Θα γίνουν άτυπες ε, συζητήσεις με τις χώρες της περιοχής που εκπροσωπούνται για να προγραμματίσουμε τη συνεδρίαση του Οκτωβρίου. Η θαλάσσια ασφάλεια θα είναι κάτι που σίγουρα θα συζητηθεί και αν δείτε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων προ 15 μέρου θα δείτε ότι υπήρξε κάποια πρόταση να έρθουμε σε επαφή με άλλες χώρες περιοχής, ευρύτερες περιοχής, με τις χώρες του κόλπου Φερρυπίν. Οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αναφέρθηκαν από κάποιου ομιλητέ. Ποια είναι η ιδέα. Θα δούμε κοινά συμφέροντα. Ποια είναι. Η ασφάλεια των θαλασσών πιθανότατα θα είναι ένας τομέας. Υπάρχει μακροσκελής κατάλογο στα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με αυτό. Και αυτό λαμβάνεται υπόψη. Για μελέτες όσον αφορά την πειρατεία και το έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα φτάνουμε στο τέλος μιας σύντομης μελέτης που δίκατσε πολύ τις ε, υπηρεσίες του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά και το έγκλημα. Ε, προσπαθεί να κάνει μια ανάλυση, να δούμε ποια στοιχεία που χρησιμοποιήσουμε για περαιτέρω επενδύσεις όσον αφορά την ασφάλεια των θαλασσών ίσως σε συνεργασία με χώρες του κόλπου, αλλά και παράκτια αστική ανάπτυξη που όπως αναφέρθηκε με τις ακτές της Ομαλίας που είναι μεγάλου μήκους σίγουρα υπάρχουν δυνατότητες. Δεν είμαι σίγουρη κατά πόσο εγώ ή το πάνελ καλύτερα θα μπορούσε να απαντήσει συγκεκριμένε ερωτήσει για εκείνου που εκπαιδεύονται και για τις άδειε για αλληλεία. Μπορώ να ελέγξω τα στοιχεία που έχουμε για τα σχετικά προγράμματα και να σε ενημερώσω. Νομίζω ότι κάλυψα τα πάντα. Αν υπάρχει κάτι που θα πείτε το όμως, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου. Ερώτηση έχω κι εγώ. προς τον πλήρχο Μαρτινούτσι απευθύνεται βασικά. Αλλά και άλλοι παριστάμενοι ε, ίσως θα θελήσουν να πούν κάτι. Στην επιχείρηση Αταλάντα, όπως είπαμε και στο Northwood, η συλλογή πληροφοριών ήταν κάτι σημαντικό. Η συλλογή πληροφοριών λοιπόν με τη συνεργασία του τομέα των ε, πλειοκτητών ε, αυτός ο παράγοντας μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτενέστερα για την επιχείρηση αυτή μετά την αλλαγή του αρχηγείου πόση από την υφιστάμενη υποδομή της επιχείρησης Αταλάντα θα αλλάξει. Μόνο το αρχηγείο ή θα υπάρχουν και άλλες συνέπειες. Άλλη ερώτηση. Όσον αφορά τις δράσεις κατά της πειρατείας και τις νομικές πτυχές. Υπάρχει ανάγκη σύναψης συμφωνιών με χώρες της περιοχής νομικού περιεχομένου, πιθανότατα. Άλλα μέλη επιθυμούν να πούν κάτι. Καλώς. Ο πλήρχος, αν έχει την καλοσύνη, ας μας ε, δώσει κάποιες πληροφορίες. Και κυρία μου και εσείς, αν θέλετε να πείτε κάτι, να αισθανθείτε ελεύθεροι ο πλήρχος Μαρτινούτσι. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να αναφερθώ σε αυτά τα δύο θέματα και επειδή εγώ ήμουν διοικητής της Αταλάντα του 2015 μπορώ να πω κάποια πράγματα. Πέρασε καιρός, πολύ καιρός, αλλά κάτι θυμάμαι ακόμα. Για, τα, για τις πληροφορίες, συλλογή πληροφοριών και μυστικές υπηρεσίες συλλέγονται οι πληροφορίες ποικιλοτρόπως. Μέσω drones, μέσω δορυφόρων, αλλά και άλλος καλός τρόπος συλλογής πληροφοριών είναι οι ανθρώπινες πηγές όπως αποκαλούμε. Στις περιπολίες με το σκάφος ερχόμαστε σε επαφή με τους ντόπιου ψαράδες επικοινωνούσαμε μέσω ασυρμάτου με όλα τα σκάφη που πέρναγαν από την περιοχή των επιχειρήσεων. Για να συλλέξουμε στοιχεία. Ποιοι είναι, πού είστε, παρακαλώ απαντήστε τους λέγαμε στον ασύρματο. Ποιο είναι το φορτίο σας. Αυτού του είδους στοιχεία θέλαμε να συλλέξουμε. Αυτά τα χρησιμοποιούσαν οι αρμόδιες δομές στο αρχηγείο, στη Βρετανία. Και στο Northwood, στο αρχηγείο, αναπτύξαμε το Κέντρο Θαλασσίων Επιχειρήσεων της, του, του Κέρατος Αφρικής. Αυτό είναι φορέας που δρά στο αρχηγείο και είναι ένα σημείο διαπαφής μεταξύ της διεθνούς ναυσιπλοείας και των στρατιωτικών στοιχείων για να γίνει συντονισμός προσπαθειών μεταξύ εμπορικής ναυτιλίας και πολεμικού ναυτικού. Και αυτό ούτω ώστε να αυξηθεί η αντοχή και η προστασία των εμπορικών πλοίων. Εμσιτσούα λέγεται αυτός ο φορέας. Θέλουμε να ανταλλάξουμε, να αναπτύξουμε την βέλτιστη πρακτική διαχείρισης. Είμαστε στην πέμπτη εκδοχή, δηλαδή να δίνουμε συμβουλές και συστάσεις στα σκάφη. Πώς να συμπεριφερθούν και πώς να πάρουν αμυντική στάση ούτω ώστε να δυσκολέψουν τη ζωή ε, των πειρατών όταν αυτοί επιτεθούν. Η MC2 επίσης προσπαθεί να συντονίσει και όλη τη διέλευση των πλοίων, δηλαδή να δίνει συμβουλές στα εμπορικά σκάφη που περνούν από τους εμπορικούς διαδρόμους, αν υπάρχει νιοπομπή που έχει οργανωθεί από διεθνείς φορείς, από τις συνδυασμένε θαλάσσιες δυνάμεις που, των οποίων ηγούνται οι ΙΠΑ να επιτρέψει αυτό το σχήμα ε, ασφαλή διέλευση των σκαφών και να δίδονται συμβουλές στην αρχή και το τέλος της διέλευσης να υπάρχει μια εξακρίβωση, ένας έλεγχος. Άρα ελέγχεται όλη η κυκλοφορία που κινείται προς δυτικά, ανατολικά, προς τον κόλπο του Άντεν και να δίνουμε συμβουλές για την ασφάλεια. Δεν υπάρχει εθνέ θαλάσσιο κέντρο διάσωσης σε αυτή τη φάση. Άρα είναι πάντα παρούσα για αυτό το σκοπό ασφαλεία στη θάλασσα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά το μέλλον, στο αρχηγείο του Northwood, όπως το είδαμε εμείς το θέμα, είναι ότι στο Ισπανικό αρχηγείο σε κοινοπραξία με τις γαλλικές αρχές προτείνουν μια ρύθμιση. Ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση των επιχειρήσεων θα είναι στα, στο Ισπανικό Αρχηγείο, στη Ρώτα. Η μεταφορά αρμοδιοτήτων του Κέντρου Θαλωσίου Μεταφορών για το κέντρο ε, της, ε, για το κέρας Αφρικής θα πάει στη Βρέστη, στη Γαλλία. Οι δύο φορείς θα πρέπει να συντονιστούν, να δημιουργήσουν κατάλληλο μηχανισμό συντονισμού για να αποδώσουν με αποτελεσματικότητα και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες στα ίδια επίπεδα όπως και στο Northwood. Θα γίνει αξιολόγηση σχετική και από πλευράς γαλλικής και από πλευράς ισπανικής. Επί του παρόντος η προσφορά τελεί υπό από την αρμόδια επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ετοιμάζεται και απόφαση του Συμβουλίου για τη μεταφορά ε, του αρχηγείου και των εξουσιών του αρχηγείου στις νέες τοποθεσίες. Δράτω με τις ευκαιρίες που αναφέρομαι στη Ρέλεξ να μιλήσω για τις νομικές πτυχές. Όταν αποφασίζεται ξεκινά μία αποστολή στρατιωτική είναι ένα ζωντανό σύστημα που πρέπει το σύστημα αυτό να τεθεί στο κατάλληλο πλαίσιο. Δεν πρόκειται μόνο μεταφοράς του ελέγχου και των διαταγών από το ένα κέντρο και στο άλλο. Αυτό προσπαθεί να το κάνει το Ρέλεξ. Και να διευθυνθούν όλες οι νομικές λεπτομέρειες και να υπάρχει και νομική βάση για να μεταφερθούν οι νομικές αρμοδιότητες ε, στη Βρέστη και στην Ισπανία. Νομίζω, λέει η Πρόεδρος, ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτό το τμήμα των συζητήσεων. Ευχαριστώ τους συγκεκριμένου προσκεκριμένους μας, τα μέλη του πάνελ που μίλησαν, που απάντησαν σε ερωτήσεις. Θα εστιαστούμε στο θέμα του κέρατος της Αφρικής αργότερα, ακόμα και κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας. Θα συναντηθούμε για μία ακόμη φορά και ίσως και πιο συχνά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. I think that Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε το επόμενο σημείο μετά από ένα λιγόλεπτο διάλειμμα για να γίνει μια ανακατάταξη εδώ στις θέσεις.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 the Λοιπόν, έχουμε την εξοχότητά της, την κυρία Μπάλφορντ, Γιαννάκα Μπάλφορντ, εκπροσωπεί την Ολλανδία. Στο PSC e και συμφωνούμε ότι ένα από τα βασικά σημεία της παρουσίασής της θα είναι το MH17, η πτήση MH17. Η πτήση λοιπόν, η οποία κα, καταρρίφθηκε πάνω από το ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας. Και τώρα έχουμε τα απορίσματα των ερευνών, πολύ ενδιαφέροντα, που θα παρουσιαστούν από την πρέσβυρα την κυρία Μπάλφορτ. Έχετε το λόγο τώρα αμέσως κυρία πρέσβυρα. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που μπορώ να έρθω εδώ και να ανταλλάξουμε απόψεις για το σημαντικό το θέμα αυτό για την Ολλανδία, της κατάρριψης της πτήσεως MH17. Ένα χρόνο είμαι εδώ τώρα αλλά για πολλούς Ολλανδούς ξέρουμε που βρισκόμαστε 17 Ιουλίου του 2014, το θυμόμαστε. Εγώ ήμουνα στην πρεσβή μας στη Ουάσιγκτον τότε και ξέρω ξεκάθαρα τι συνέβη και γνωρίζω και θυμάμαι ότι ο τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ομπάμα, επισκέφθηκε την πρεσβεία μας για να μα συλληπιθεί και να γράψει συλληπιτήρια στο βιβλίο συλληπιτηρίων της πρεσβείας. Μετά από αυτό συζητήσαμε εκτενώς με τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών το θέμα της πτήσεως MH17 και από την αρχή ήμασταν ξεκάθαροι. Είπαμε ότι χρειάζεται μια εσβάθος έρευνα για εκείνους που δεν γνωρίζουν ακριβώς τι συνέβη ήταν ένα αεροσκάφος της Malaysian Airlines, των Μαλαισιανών αερογραμμών, που καρτερίφθη πάνω από τον ενέργειο χώρο στις 17 Ιουλίου του 2014 είχε 298 επιβάτες από αυτούς 198 ήταν Ολλανδοί πολίτες Διεξήχθη έρευνα από το Ολλανδικό Συμβούλιο Ασφαλείας με πληροφορίες που έδωσε η Αυστραλία, το Βέλγιο, η Μαλαισία, η Ρωσική Ομοσπονδία, η Ουκρανία και οι Ηνωμένε Πολιτείε και η σχετική έκθεση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ολλανδικού έδειξε ότι καταρρίφθηκε με πύραυλο που ε, ε, εκτοξεύθηκε από την βάση Μπουκ από το έδαφος της Ουκρανίας. Η περιοχή ήταν υπό τον έλεγχο των αποσχιστικών δυνάμεων, περαιτέρω έρευνες από την μεικτή ερευνητική ομάδα διεξήχθη. Αποτελείται αυτή η ομάδα από την Ολλανδία, την Αυστραλία, το Βέλγιο, τη Μαλαισία και την Ουκρανία και συνεπέραν η ομάδα ότι ακριβής φύσης του όπλου που χρησιμοποιήθηκε που εκτοξεύτηκε από τη βάση Μπουκ ήρθε από τη Ρωσική Ομοσπονδία στην Ουκρανία και επέστρεψε μετά ο εκτοξευτήρας αφού έγινε η επίθεση κατά της MH17. Και αυτή η έρευνα δημοσιοποιήθηκε στις 24 Μαΐου. Η κοινή ερευνητική ομάδα συνεπέρανε ότι ο εκτοξευτήρας Μπουκ ανήκε στη Ρωσική Ομοσπονδία στο 53ο Σύνταγμα Αντιεροπορικού Πολέμου. Στις 25 Μαΐου η Αυστραλία και το Βασίλειο της Ολλανδίας φρονούν ότι η Ρωσική Ομοσπονδία μέσω του ρόλου που έπαιξε στην κατάρριψη του MH17 τον Ιούλιο του 2017 παραβίασε διάφορες υποχρεώσεις του διεθνούς δικαίου και η Ολλανδία και ε, η Αυστραλία θεώρησαν ότι η παραβίαση του διεθνούς δικαίου αποτέλεσε ε, κατακριτέα αξιόπινη ε, πράξη και φέρει την ευθύνη η Ρωσική Ομοσπονδία. Παρουσιάσαμε ένα σημείωμα, το υποβάλαμε στη Ρωσική Ομοσπονδία, ούτως ώστε να θέσουμε τη Ρωσική Ομοσπονδία πρώτων ευθυνών της και είπαμε ότι η ευθύνη έχει νομικές συνέπειες για τη Ρωσική Ομοσπονδία και ζητήσαμε από τη Ρωσική Ομοσπονδία να αποδεχθεί πλήρως τις ευθύνες της για τις διεθνείς αυτές πράξεις να δώσει στην Αυστραλία και στο Βασίλειο της Ολλανδίας τις κατάλληλες διαβεβαιώσεις και εγγύσεις για μια επανάληψη αυτών των διεθνών αξιόπινων πράξεων και να δώσει στην Ολλανδία, και στην Αυστραλία πλήρες αποζημιώσεις που απορρέουν από αυτές τις ε, πράξεις. Είναι ένα ξεχωριστό μονοπάτι που η Ολλανδία και η Αυστραλία ακολούθησαν για να θέσουν τη Ρωσική Ομοσπονδία πρώτων ευθυνών της. Εν τω μεταξύ, η έρευνα της μικτής ε, συγγνώμη, ε, ερευνητικής ομάδας συνεχίζεται ε, και υπάρχει και νομική διαδρομή που θα ακολουθηθεί και δικαστική στην Ολλανδία. Αυτό είναι ένα άλλο βήμα που από κοινού η Ολλανδία και η Αυστραλία ακολουθούν για να θέσουν τη Ρωσική Ομοσπονδία πρώτων ευθυνών της. Εν συντομία, αυτά συνέβησαν τον Μάιο και αυτή ήταν η απόφαση της Ολλανδικής κυβερνήσεως να τεθεί η Ρωσική Ομοσπονδία πρώτων ευθυνών της. Θέλουμε να δούμε ποιες θα είναι οι πράξεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας, παρακολουθούμε, έγιναν συζητήσεις επ' αυτού στο κοινοβούλιο μας, αυτό είναι ένα νομικό βήμα το οποίο κάναμε για να θέσουμε τη Ρωσική Ομοσπονδία πρώτων ευθυνών της και για την ώρα αυτό είναι το βήμα που κάνουμε και όχι άλλα πέρα τη συνέχιση των ερευνών που ελπίζουμε ότι τελικά θα, ε, μέσω της έρευνας θα βρούμε στοιχεία για τα υπεύθυνα άτομα που θα προσαχθούν, θέλουμε να προσαχθούν στη δικαιοσύνη. Θα σταματήσω εδώ, ούτω ώστε να δώσω τη δυνατότητα να υποβληθούν ερωτήσει και να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσει από αυτού. Μάλιστα, σα ευχαριστούμε. Ο κύριος Γκάλερ, ευχαριστώ πολύ. Εγώ προσωπικά θυμάμαι που ήμουν εκείνη την μέρα και ώρα όταν συνέβη. Ήταν πέμπτη απόγευμα, ήμουν σπίτι και θυμάμαι ότι κοιτούσα στο διαδίκτυο τα νέα. Διάβαζα μια ρωσική εφημερίδα στα γερμανικά. Όταν διάβασα για την κατάρριψη του αεροσκάφους, μάλιστα ε, αναφερόταν σαν ουκρανικό της πολεμικής αεροπορίας. Έλεγξα κατόπιν την είδηση και στο αγγλικά και συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν καθόλου ουκρανικό πολεμικό αεροσκάφος, αλλά το MH17, μια πτήση της ε, πολιτικής αεροπορίας ε, της Malaysian Airlines. Εξαφανίστηκε μάλιστα η είδηση κατόπιν και από το αγγλικό και από το γερμανικό ε, τύπο. Και φυσικά αυτό που συνέβη αργότερα είναι να μην έχουμε πληροφορίες ακριβείς. Η διαδικασία πήρε πάρα πολύ χρόνο, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να φτάσουν κάποια στοιχεία και φυσικά σήμερα ξέρουμε ότι υπήρξαν και συγκεκριμένα άτομα που έδωσαν την εντολή για να γίνει όλη αυτή η επιχείρηση κατά του αεροσκάφους. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχουν αποδείξεις σήμερα ατράνταχτες για το ποιος έδωσε την εντολή και από πού προέρχεται η επίθεση αυτή κατά του αεροσκάφους. Θα ήθελα να μου πείτε αν υπάρχει σήμερα συγκεκριμένη πρόθεση να γίνει μια διαμαρτυρία, ένα επίσημο διάβημα κατά των ρωσικών αρχών. Ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για πράξη πολέμου, αλλά η ρωσική κυβέρνηση, η ρωσική ομοσπονδία βρίσκεται πίσω από αυτήν την πράξη αποσταθεροποίησης της Ουκρανίας και διαπιστώνουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να φύγει ένας τέτοιος ε, εκτοξευτήρας και πύραυλος να περάσει τα σύνορα, να φύγει από τη Ρωσία, να πάει στην Ουκρανία και να εκτοσκευθεί χωρίς να υπάρχει ρητή άδεια και εντολή από μέρους των ρωσικών αρχών. Αυτό κανείς, κανένας ε, στρατιώτης Ρώσος δεν θα αναλάμβανε αυτή την ευθύνη μόνος του. Θεωρώ λοιπόν ότι ίσως υπάρχει σήμερα η πολιτική συγκυρία να χρησιμοποιήσουμε αυτή την υπόθεση άσχετα από οικονομικές αν θέλετε κυρώσεις και αντίπεινα. Χρειάζεται μία σαφής καταδίκη και από πολιτικής απόψεως πιστεύω ότι πρέπει να σταλεί ένα συγκεκριμένο μήνυμα, να ληφθούν πολιτικά μέτρα τα οποία να είναι αποτελεσματικά. Δεν είναι δυνατόν στον 21ο αιώνα στην Ευρώπη να λύνονται τα θέματα με τις γειτονικέ χώρες με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ πολύ, κ. Φωνζουλίκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάποια από αυτά που ήθελα να πω τα είπε ο κύριος Γκάλερ ο συνάδελφος. Θέλω να ρωτήσω την πρέσβη πόσο καιρό θα περιμένουμε μέχρι να δοθεί απάντηση από τη Ρωσική Ομοσπονδία και αν δεν σας δοθεί καμία απόφαση τι προτίθεστε να κάνετε από νομικής απόψεως τι μπορείτε να κάνετε επίσης τι κάνει η Μαλαισία, η Malaysian Airlines. Δεν ζητούν κάποια αποζημίωση ή τουλάχιστον αναγνώριση αυτού του τρομακτικού, φρικιαστικού, αν θέλετε, γεγονότος που ουσιαστικά είναι εχθροπραξία και η επίθεση κατά ενός ε, Τέτοιο αεροσκάφο είναι κάτι που δεν μπορεί να περάσει ατιμόρυτο. Κύριε Χάμ. ευχαριστώ πολύ την Ολλανδία και όλες τις άλλες χώρες που συμμετείχαν σε αυτή τη διερευνητική ε, ομάδα. Παρακολούθησα τη συνέντευξη τύπου από την αρχή μέχρι το τέλος, όταν, όταν παρουσιάσετε συγγνώμη τα αποτελέσματα αυτής της, όπως τη λέτε, ε, τελικά τα προσωρινής έκθεσης συμπερασμάτων. Έτσι όπως παρουσιάστηκε αυτή η έκθεση και τα συμπεράσματα, όλοι, αυτοί τουλάχιστον που το έχουν ε, ακούσει και δει, θα πρέπει να το διαβάσουν πολύ προσεκτικά πριν συζητήσουμε για τις πολιτικές και νομικές συνέπειες. Πιστεύω ότι χωρίς τη δική σας μαρτυρία, χωρίς τα δικά σας συμπεράσματα, θα είναι πολύ δύσκολο για συναδέλφους εδώ να συζητήσουν τις συνέπειες, τις πιθανές συνέπειες. Εγώ Φυσικά και πιστεύω ότι από την πρώτη μέρα υπάρχει ευθύνη ρωσική. Ήμουν στο Χάκεπ θυμάμαι και είδα τις αρχές να προσπαθούν να συνεργαστούν με τις αρχές ε, στον Ντόνιετς και μπορώ να σας πω πως από τη μία στιγμή στην άλλη οι αρχές των Ντόνιετς διέκοψαν κάθε επαφή με τις Ουκρανικές ε, αρχές. Είδαμε λοιπόν καθυστέρηση και στις έρευνες και στις εποστολές διάσωσης. Πέρασαν ε, βδομάδες και η διερεύνηση της υπόθεσης με στο καλοκαίρι, φρικτές συνθήκες, ζέστη και όλοι όσοι συμμετείχαν στην έρευνα εκείνο το καλοκαίρι και τα συμπεράσματα στα οποία έχουν φτάσει όλοι συμφωνούν. Αναρωτιέμαι λοιπόν ποιο θα είναι το επόμενο βήμα, τι προτίθεστε να κάνετε όσον αφορά τις ευθύνες της Ρωσίας. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξουν διπλωματικές συνέπειες, νέες κυρώσεις, προσφυγή στη δικαιοσύνη. Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική κατά της Ρωσίας. Πώς μπορούμε να εμπλακούμε. Είναι περίεργο να υπάρχει αυτή η έρευνα, να υπάρχουν συμπεράσματα, αλλά δεν υπάρχουν συνέπειες. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση, λέει Πρόεδρος. Θα ήθελα να αποτίσω φοροτιμής προς την Ολλανδία, την κυβέρνηση, την αυτού τη βασίλισσα, τους πολίτες της Ολλανδίας όσον αφορά αυτή την καταστροφή, αυτό το έγκλημα εμείς στην Πολωνία το παρακολουθούμε στενά και σκέφτομαι και κάποιο άλλο τέτοιο περιστατικό και καταστροφή που συνέβη στη χώρα μας. Ποια είναι λοιπόν τα μέτρα που προτίθεστε να λάβετε Μπορείτε να μας πείτε ποιοι είναι οι εταίροι τη συνεργασία έχετε μαζί τους, πώς κατανεμήθηκε μέχρι τώρα, πώς έχει κατανεμηθεί μέχρι τώρα, συγγνώμη, η ε, τεχνική υποστήριξη, η βοήθεια, η διερεύνηση της υπόθεσης όσον αφορά τη χρήση της βάσης του book και όσον αφορά την εμπλοκή των ε, δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Θέλω να κάνω μία παρατήρηση. Μετά την ε, παράνομη προσάρτηση της Κρυμαίας συνέβη αυτό το περιστατικό με την πτήση MH17. Και βλέπουμε ποια είναι η στάση της Ρωσίας γενικότερα έναντι της Δύσης. Τον Απρίλιο του 10 η στάση της Ρωσίας ήταν εντελώς διαφορετική. Το περιβάλλον ε, ήταν εντελώς διαφορετικό και όλος ο δυτικός ε, δημοκρατικός κόσμος ήθελε να υπάρξει πιο σοβαρός διάλογος, πιο βαθύς διάλογος με την Ρωσία. Βλέπουμε ότι σήμερα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, έχουν αλλάξει. Και από την αρχή εμείς ε, γνωρίζαμε ότι αυτή η βίαιη πράξη της Ρωσίας ε, ήταν κάτι που γνωρίζαμε ότι προέρχεται από τη Ρωσία και μάλιστα μας κορόιδευαν τότε όταν το λέγαμε. Και πραγματικά αυτή η εκστρατεία παραπληροφόρησης αν θέλετε που ουσιαστικά ακολούθησε αυτή την ιστορία με την πτήση MH17 είναι κάτι που προσπάθησε να αντικρούσει η Ολλανδία. Αλλά πρόκειται για παρόμοιες, αν θέλετε, ε, επιθέσεις και λίγα λεπτά ουσιαστικά μετά την τραγωδία που έλεγε χώρα στη χώρα μας, ακούσαμε ότι ο πιλότος του εν λόγω πολωνικού αεροσκάφους ήταν ανίκανος, ήταν μεθυσμένος, ήταν ε, δικό του φάλμα. Ευχαριστώ πολύ και σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ και θα προσπαθήσω να απαντήσω καταρχήν στον κύριο Γκάλερ όσον αφορά τα πολιτικά βήματα που θέλουμε να αναλάβουμε. Ήδη στις 9 Μαρτίου στείλαμε μια επιστολή στο κοινοβούλιο μας λέγοντας ότι υπάρχει κρατική ευθύνη. Από την ημέρα που καταρρίφθηκε αυτό το αεροσκάφος θέλουμε και το έχουμε ανακοινώσει να βρεθεί η αλήθεια, να συνεχιστεί η έρευνα και να υπάρξει λογοδοσία των υπευθύνων. Συνεχίζουμε σε αυτή τη γραμμή και επιθυμούμε να ληφθεί απόφαση πρώτον όσον αφορά την ευθύνη από μέρους αυτού του κράτους και να συνεχιστούν οι έρευνες, όπως είπε και η κυρία Χάρμς. Δεν πρόκειται για μια τελική έκθεση και τελικά συμπεράσματα. Η έρευνα συνεχίζεται και συλλέγονται στοιχεία. Θέλουμε να προσαχθούν οι υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη. Αυτή είναι η αποστολή του εισαγγελέα από την Ολλανδία. Τι μπορεί να κάνει, ρωτάτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε πολλά στηρίζοντας όλα τα βήματα της εν λόγω διαδικασίας στην ε, διαρεύνηση της υπόθεσης και τα νέα συμπεράσματα αυτής της ε, μικτής ε, διερευνητικής επιτροπής έχουν στηριχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητήσαμε από όλους τους εταίρους μας να στηρίξουν τα αποτελέσματα δημοσίως, κάνοντας ε, δημόσιες ανακοινώσεις. Ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει την απόφαση της κυβέρνησης της Ολλανδίας και είμαστε ευγνώμονες γιατί υπήρξε δήλωση των 28 την ίδια μέρα που επαναλαμβάνει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από την 2166 ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας και το γεγονός ότι αυτή η κοινή διερευνητική επιστολή, ε, επιτροπή έχει διεξάγει μια ανεξάρτητη και αμερόληπτη έρευνα κατονομάσαμε και την Ρωσία ως υπεύθυνη. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίζει να στηρίζει το αίτημά μας να δεχτεί δηλαδή η Ρωσία την ευθύνη της και να δοθούν περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες τα οποία ζητούμε εδώ και καιρό από τις ρωσικές αρχές. Συνεχίζουμε λοιπόν να ζητούμε τη στήριξη όλων. Αυτά είναι τα βήματα που θέλουμε να αναλάβουμε, θέλουμε να συνεχίσουμε. Κύριε Φανσολίκα, όσον αφορά περαιτέρω δράση, θα συνεχίσουμε σε αυτή τη γραμμή και στοχεύουμε να ενισχύσουμε αυτή μας τη θέση. Η μεικτή διαπραγματευτική ομάδα συνεχίζει το έργο της συλλογής στοιχείων μέχρι να προσαχθούν οι υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη. Προς το παρόν, τα δύο βήματα που έχουμε αποφασίσει είναι αυτά τα δύο που σας περιέγραψα. Αργότερα θα υπάρξουν και άλλα βήματα, δεν ξέρουμε ακριβώς πια. Προς το παρόν έχουμε αυτά τα δύο και θέλουμε πραγματικά να οδηγήσουμε τη Ρωσία να συνεργαστεί, να απαντήσει και ζητούμε από όλους να μας στηρίξουν στο δρόμο αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας και Συνεργαζόμαστε και με την κυβέρνηση της Μαλαισίας. Η Μικτή Διερευνητική Επιτροπή, στην οποία συνεργάζεται και η Μαλαισία. Κυρία Χάρμς, να απαντήσω σε αυτό που με ρωτήσατε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή για τους Ουκρανούς να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους. Ήταν εξαιρετικά χρήσιμη, συνεργάσιμη από την αρχή, αλλά καταλαβαίνετε ότι υπάρχει θέμα και με την ε, νομική ασφάλεια όλοι όσοι παραδείγματο χάρη έχουν ε, καταθέσει σαν μάρτυρες, δεν ξέρουμε τι μπορεί να του συμβεί. Είναι δύσκολη η επικοινωνία, παρόλα αυτά πάρα πολλοί άνθρωποι στην Ουκρανία μας στήριξαν, αλλά και διεθνείς ε, εταίροι, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μαζέψουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Κυρία Φωτίγα, ναι, από την αρχή η έρευνα αυτή ήταν και τεκμηριωμένη και επιστημονική, αλλά και αμερόληπτη. Η κυβέρνηση της Ολλανδίας δεν γνωρίζει από την αρχή το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας. Ανήκουμε στην ομάδα και συνεργαζόμαστε στενά με τους εισαγγελείς, οι οποίοι συνεχίζουν την δουλειά τους. Δύσκολη όμως ήταν η όλη διαδικασία. Συνεχίζουμε να βρίσκουμε στοιχεία αξίζει τον κόπο να τα γνωρίζουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και είναι σαφές ότι η κυβέρνηση της Αυστραλίας και η κυβέρνηση της Ολλανδίας ε, ρίχνουν ευθύνες και κατανομάζουν την Ομοσπονδία της Ρωσίας. Είμαστε πεπισμένοι ότι θα πρέπει να αφήσουμε τους εισαγγελείς να δουλέψουν αμερόληπτα και σοβαρά. Μία συμπληρωματική ερώτηση έχω όσον αφορά τις πηγές στοιχείων για μας, για το γενικό ε, κοινό. Αυτή η ανακοίνωση που κάνατε όσον αφορά τα στοιχεία Είμαι 100% πεπισμένο σήμερα ότι οι Αμερικάνοι φίλοι γνώριζαν πολύ καλά τι συμβαίνει στην περιοχή μέσω δορυφορικής παρακολούθησης και σε πραγματικό χρόνο. Ξέρουν πολύ καλά από πού έφυγε ο πύραυλος. Σας έδωσαν πληροφορίες άμεσα οι αμερικανικές πηγές. Δεύτερον, δεύτερη ερώτηση οι Ρώσοι λένε ότι δεν ε, μπόρεσαν να συμμετάσχουν σε αυτή την κοινή διερευνητική ομάδα. Καταλαβαίνω γιατί, δεν χρειάζεται να μου εξηγήσετε, αλλά ποια είναι τα επιχειρήματα που τους αντιτάξατε για την μη συμμετοχή τους σε αυτή την ε, μεικτή ομάδα. Κυρία Ρεμπέκα Περισσότερο μια παρατήρηση παρά ερώτημα. Όσο μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάσετε τα βρήματα της έρευνας για πολλούς λόγους ε, και για τις οικογένειες των θυμάτων και τους Ουκρανούς θεωρώ ότι ήταν μια πολύ σημαντική ημέρα. Αλλά Ταυτόχρονα με εντυπωσιάζει το γεγονό ότι στην δισογραφία της Γερμανίας, στο πρώτο κανάλι ή στο, στα δημόσια, στις δημόσια ραδιοφωνικές εκπομπές δεν χρησιμοποίησαν ποτέ τη διατύπωση κατάρριψη. Δηλαδή παρέμεινε ανοιχτό τι ακριβώς είχε συμβεί παρά τις δημοσιεύσεις που κάνατε. Και νομίζω ότι αυτό ε, μας δίνει κάποια στοιχεία σχέση με τον πόλεμο ενημέρωσης ε, και μας παρέχει αποχρόντως λόγους να συνεχίσουμε να τα ευρήματα. δεν πρόκειται μια στιγμή όπου κανείς ε, που ενδιαφέρεται κάπως παρακολουθεί και την επομένη βρισκόμαστε στον κόσμο αυτών της ειδησογραφίας όπου τα νέα είναι ισορροπημένα όπως λένε εντό εισαγωγικών και από τις δύο πλευρές. Εδώ όμως δεν πρόκειται για ισορροπία, αλλά για παρουσίαση δεδομένων πραγματικών γεγονότων. Και ιδιαίτερα αυτό που είπατε, η παρουσίαση των πραγματικών γεγονότων, είναι ο λόγος για τον οποίο είμαστε πολύ προσεκτικοί στην παρουσίαση αυτή. Παρουσιάσουμε πραγματικά γεγονότα και δίνουμε έμφαση στην αμεροληψία της ε, ερευνητικής ομάδας. Η κοινή ερευνητική ομάδα αποτελείται από ομάδες οι οποίες ε, επηρεάστηκαν από την κατάρριψη του αεροσκάφους το οποίο είχε πάρα πολλές απώλειες ε, ε, η Μαλαισία και η Ουκρανία σαφώς επλήγησαν. Ρωτήσαμε κατά επανάληψη, ζητήσαμε τη Ρωσική Ομοσπονδία να συνεργαστεί με την ερευνητική ομάδα. Συνεχώς τους ζητούσαμε πληροφορίες και τους καλέσαμε να συνεργαστούν κατ' επανάληψη σε διάφορες περιστάσεις ακριβώς όπως ε, συνεργαστήκαμε με τις ΙΠΑ για την παροχή πληροφοριών αλλά πολύ προσεκτικά γιατί η κοινή ερευνητική ομάδα ε, συστάθηκε για να εργαστεί ξεχωριστά από την κυβέρνηση της Ολλανδίας. Υπήρξε λοιπόν επίσημο αίτημα εκ μέρους τη Ολλανδική κυβέρνησης προ τη Ρωσική κυβέρνηση να συνεργαστεί, αλλά επίσης υπήρξαν και άλλα ε, νομικά αιτήματα συνεργασία προ τη Ρωσική Ομοσπονδία. Βεβαίω συνεργαστήκαμε επίση και με τι Αμερικανικές αρχές. Και ελέγξαμε όλες τις πληροφορίες Και ε, κάναμε μια προσεκτική εξέταση όλων των πληροφοριών. Γι' αυτό όλα αυτά ε, ε, ε κράτησαν πολύ χρόνο και δεν είναι εύκολο να το εξηγήσουμε. όπως λέει η κυρία Χάρμς, για τον πόλεμο ενημέρωσης και το γεγονό ότι οι δεν βασίζονται πάντα σε πραγματικά γεγονότα. Αλλά εμεί θέλαμε να εξασφαλίσουμε ότι πρόκειται για μια αντικειμενική αμερόληπτη έρευνα και όλα τα στοιχεία ε, τα οποία διοχετεύθηκαν προς την ε, εισαγγελία ελέγχθηκαν ως προς την ακρίβειά τους. Πόσο σημαντικός ήταν ε, ο έλεγχος των ε, τμήματων του ε, αεροσκάφους. Έγινε ανα κατασκευή ολόκληρου του αεροσκάφους. Ε, ήταν πολύ σημαντικό αυτό το, θέμα και συνεργαστήκαμε με διάφορους ε, εταίρους, με διάφορες χώρες για τις έρευνες στα εργαστήρια γιατί ορισμένες χώρες είχαν μια καλύτερη εμπειρία και συνεργαστήκαμε μαζί τους. Αλλά όσο για τον ακριβή τρόπο που έγινε δεν μπορώ να σας πω. Συνάδελφοι, παρακαλώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την αυτού εξοχότητα για την πολύ ενδιαφέρουσα και ειλικρινή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για μια απόθεση εξαιρετικά τραυματική για όλη την Ολλανδική κοινωνία. Εξ αρχής ε, σταθήκαμε στο πλευρό σας και υπήρξαμε υποστηρικτικοί. Σας ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία. Okay, colleagues. Uh, Συνάδελφοι, ε, εδώ ε, ολοκληρώνεται η συνεδρίαση. Η προσεχή συνεδρίαση είναι στις 6 Σεπτεμβρίου. Στις 6 το απόγευμα έχουμε ένα διευρυμένο προεδρείο με σημαντικές αποφάσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Γραμματεία και όλους σας για τη συμμετοχή σας. Βεβαίως και τους διερμηνείς για το εξαιρετικά σημαντικό τους και εξαίρετο έργο. Ευχαριστώ.